Ehm, λοιπόν, γεια σας. Ε, θεωρούμε δεδομένη την υιοθέτηση της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Συζήτηση για την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρίση στον τομέα της αλληλείας λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάντεκ. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία έδρα έχει μόνο και αυτό είναι, ε, βρίσκεται στο Στρασβούργο. Από το Φεβρουάριο του 2011 η τιμή του πετρελαίου διαρκώς αυξάνεται. Έχει υπερβεί και ε, τα 100 δολάρια πλέον. Οπότε οι σε όλες τις παράκτες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την ε, σημαντική αυτή αύξηση του, της τιμής του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν κανέναν αυτά που λέω. Ενημερώστε με. Αν δε, πάλι δεν σας ενδιαφέρει να μου το πείτε. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα περιμένω για να αναχωρήσουν όσοι να αναχωρήσουν. Συνάδελφοι. Όποιος θέλει να φύγει παρακαλώ να το κάνει αμέσως και χωρίς να κάνει θόρυβο, χωρίς να καθυστερεί και να στέκεται να συζητά στους διαδρόμους. Λοιπόν, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στον κύριο Καντέκ να πάρει το λόγο χωρίς να ενοχλείται. Κύριε Καντέκ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, σας ξαναρχίζουμε τον χρόνο από την αρχή, κύριε Καντέκ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα επαναλάβω, ζητώ συγγνώμη, μία έδρα έχει το Κοινοβούλιο και αυτή βρίσκεται στο Στρασβούργο. Ε, από το Φεβρουάριο του 2011 αυξάνεται διαρκώ η τιμή του πετρελαίου και υπερεύει και τα 100 δολάρια πρόσφατα. Οι αλλοί σε όλε τι περιοχές περιοχέ πλήττονται πάρα πολύ από την σημαντική αυτή αύξηση τη τιμή ε, του πετρελαίου. Ε, έχουν απογειωθεί οι τιμές ε, εκμετάλλευσης, ε, κυρίως για την ερασιτεχνική αλία, λόγω της σημαντικής αύξησης τιμής του πετρελαίου και οι ερασιτέχνες αλίες εξαρτώνται φυσικά από την τιμή του πετρελαίου. Οι επαγγελματίε εκδηλώνουν την ανησυχία τους λόγω της σημαντικής αυτής αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις παρά την υπέρμετρη αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων. Ζητώ λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη ενδεχομένως να επικουρήσουν ε, τον, κλάδο αυτό για να ε, συνεχίσουν να λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις χωρίς όμως να έχουμε στρέβλος του ανταγωνισμό, Οπότε ζητώ αύξηση από 30.000 σε 60.000 του ανωτάτου ορίου de minimis ενίσχυσης για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν επιβαρύνει αυτό τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτές οι ενισχύσεις χορηγούνται από τα κράτη-μέλη προς τις ελληνικές εκμεταλλεύσεις στο μέτρο που δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Ζητώ λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία από πλευρά των κρατών μελών. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει εις ε, το αίτημά μα και να κατανοήσει τι ε, ανησυχίε ενό ε, κλάδου που πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί η αλία. Τι σημαίνει η αλία, άντρε και γυναίκε που χρειάζονται ένα αξιοπρεπέ εισόδημα. Πρέπει να το στηρίξουμε κυρίω λόγω των εισαγωγών των ψαριών και των προϊόντων ηχθειοκαλλιέργεια από τρίτε χώρε. Γίνεται, πιο ευπαθή ο κλάδο. Δεν είναι θέμα μόνο οικονομικού κέρδους. Είναι προ συμφέρον όλων να διατηρηθεί αυτή η δραστηριότητα για, τι για τις χωροταξικές ε, των παρακτήων περιοχών και για να στηρίξουμε την απασχόληση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό κλάδο, σε αυτές τις παράκτιες περιοχές. Παρόλα. Ευχαριστώ κύριε Κάντεκ και τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπέλντερε και εκείνο για δύο λεπτά. ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. η κατάσταση στον τομέα της αλίας είναι πραγματικά ανησυχητική. Οι τιμέ των καυσίμων έχουν αυξηθεί και οι τιμέ των αλλιευμάτων βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο ιστορικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ σε σχέση με την αλία να λάβουμε υπόψη την κατάσταση τη αλίας και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν την Ολλανδία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη γλώσσα. Εδώ και χρόνια υπήρχε έλλειψη και τα νέα αλλιεύματα έχουν τα όμως ε, πρέπει να ασχοληθούμε και με τη γλώσσα και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή τη γλώσσα και να μην εισάγουμε πλέον φθηνά, υποκατάστατα φθηνά αλλιεύματα. Αυτό σημαίνει ότι η εντόπια γλώσσα θα πρέπει να μπορεί να πωλείται και να διατίθεται στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν να απολέσουν ακόμα περισσότερο ε, οι τιμές ε, των αλευμάτων αυτών, να πέσουν ακόμα πιο χαμηλά. Και πρέπει να δούμε ότι αν δεν διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των αλλιέων δεν θα υπάρχει αυτό το αλεύμα στην αγορά. Εδώ πρέπει άμεσα να δράσουμε. Και παρακαλώ λοιπόν να, να ληφθεί υπόψη αυτό και να είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου. Ε, ευχαριστώ. Είδα κάποιο να ε, μου ζητούσε το λόγο και νόμιζα πω ήταν για το ΚΑΤΣΔΙΑΕ. Αντίθετα, ήθελα να κάνει υπερώτηση στον κύριο Κάντεκ. Ποιο ε, θα θέλατε τώρα να υποβάλλετε την ερώτηση, Γιατί είναι εδώ τώρα ο κύριο Κάντεκ. Να δούμε αν δέχεται την ερώτηση. Ναι, λέει. Ωραία, ο συνάδελφο λοιπόν έχει το λόγο. Um, Πρόεδρε, θα είχα μια ερώτηση προς τον συνάδελφο Καρτέκ σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν, σε σχέση με την μία και μοναδική έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε συνάδελφε, ίσως θα προσέξατε ότι το Κοινοβούλιο καμιά φορά συνεδριάζει και στις Βρυξέλλες και ίσως θα προσέξατε ότι και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν ε, στις Βρυξέλλες και ότι υπάρχει και έδρα στο Λουξεμβούργο. Θα ήθελα να το λάβετε υπόψη αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Κάντεκ. Ε, θέλησα μόνο να υπενθυμίσω ότι οι συνθήκες είναι σαφέστατες για αυτό το σημείο. Η έδρα του Κοινοβουλίου ε, όπου βρισκόμαστε σήμερα και θα βρισκόμαστε για ολόκληρη τη βδομάδα βρίσκεται στο Στρασβούργο και μόνο. Προφανέστατα εργαζόμαστε στο, στις Βρυξέλλες δύο εβδομάδες το μήνα όπως και εσείς εκεί είμαι. Ωραία τα περνάω και εργάζομαι σκληρά. Αλλά η έδρα είναι εδώ στο Στρασβούργο και έτσι πρέπει να παραμείνουν τα πράγματα. Ε, Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τους ε, συνσυντάκτες. Ε, Μπρίτα Ρέμερς για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαρκής αύξηση των καυσίμων δημιουργεί σε πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια επιπρόσθετη επιβάρυνση, ένα πρόσθετο βάρος Ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι αλληλείς υφίστανται τα πάνδυνα από αυτή την αύξηση των καυσίμων, διότι τις πρόσθετες αυτές δαπάνες, τα πρόσθετα κόστη δεν μπορούν να τα αντισταθμίσουν με καλύτερες τιμές για τα αλλιεύματα. Η σημερινή κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και στην Εγγύης Ανατολή έχει ακόμα επιδεινώσει την κατάσταση, την έχει επιτείνει ακόμα πιο πολύ. Γι' αυτό πρέπει να δούμε Ποιε είναι οι επιπτώσει τη αύξηση των τιμών των καυσίμων στην οικονομία και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιοι τομεί είναι εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους και πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα καθεστώς στήριξης χωρίς να δημιουργηθούν στευλώσεις στον ανταγωνισμό όμως. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτή την κατάσταση και τις δυνατότητες. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Αλία ώστε και η ανεξαρτησία μας από, σε σχέση με εισαγωγές από, εισαγωγές από τρίτες χώρες να μην ε, διακυβευτεί. Βρισκόμαστε μπροστά στη μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Αυτό ιδιαίτερα μας υποχρεώνει σε αυτό το θέμα να είμαστε πραγματικά συνετοί και σόφρονες, να μην βιαστούμε υπερβολικά στην αντίδρασή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ούλρικ στη για δύο μισή λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Αλία βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Οι συνάδελφοι το επεσήμαναν πιο πριν. Αλείς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παραπονούνται για τη μείωση των εισοδημάτων τους που είναι και που μπορεί να απειλήσει την επιβίωσή τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί όμως μειώνονται τα εισοδήματα των αλλιέων μας. Για μένα υπάρχουν τρεις λόγοι γι' αυτό. Μείωση των αλλιευμάτων, συρρήκνωση των αλλιευμάτων, γενική μείωση των τιμών. Ακριβώς εκεί όπου είναι υγιή τα αλλιεύματα και που είναι μεγάλη προσφορά. Και τρίτον, και περί αυτού πρόκειται σήμερα, μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας για τους αλλιείς όσον αφορά τις αυξημένες τιμές καυσίμων. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλούνται οι πολιτικοί πολιτικοί να δράσουν εδώ. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε. Το τονίζω. Τονίζω ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Η πρόταση ψηφίσματο των συντηρητικών υπόσχεται περισσότερα από όσα μπορούμε να κάνουμε. Ζητεί μια αύξηση της, ε, του καθεστώτος στήριξης de minimis κατά 100% από 30 ε, σε 60 χιλιάδες ευρώ. Όμως ε, οι επιδοτήσεις για τα καύσιμα είναι κάτι που δεν μπορούν να αντέξουν πολλά κράτη-μέλη, δεν μπορούν να υπομισθούν τέτοια επιβάρυνση. Και έτσι δεν θα βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι αλλοίς, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αλλοίς. Κατά τα άλλα θα παραμείνουν και τα άλλα προβλήματα. Πρώτον, η υπερα, υπεραλίευση που θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Και δεύτερον, τα προβλήματα της ε, αλλίας και των αλλιευμάτων δεν θα επιληθούν. Όσον αφορά εδώ του Αλλή βλέπω ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας, παρότι πληρώνει 50% συγχρηματοδοτώντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να αλλάξει κάτι, κατεπηγόντω για τα υπέρ των συμφερόντων των Αλλιών. Συνάδελφοι, μέχρι την Πέμπτη ας κάνουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση και από κοινού με συνετό τρόπο, με λιγότερες διακηρύξεις, ας εργαστούμε υπέρ των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των αλλιέων. Μας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ο Ρόντουστ. Και τώρα η κυρία Ισαμπέλα Λοβέν. Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Καντέκ, που μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το τόσο θεμελιώδες ζήτημα. Ε, πρώτον, όταν μιλάμε για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, υπάρχουν ουσιαστικά δύο κλάδοι που δεν φορολογούνται με ενεργειακούς φόρους ε, η ναυτιλία και η αεροναυτιλία και το ίδιο ισχύει και για την αλία. Οπότε αναλογικός πως σε σχέση με τους υπολείπους κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται λιγότερο η αλία σε σχέση με άλλου κλάδους από την αύξηση της τιμής των καυσίνων επειδή εξαιρούνται από τις φορολογίες. Οπότε πρόκειται για μια και καλυμμένη επιδότηση η οποία έχει ήδη συμβάλει στη συνέχιση ε, της υπερεκμετάλλευση των εξαντλημένων αλλιευτικών αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Αλία τώρα τα τμήματα της αγοράς ε, που καταναλώνουν περισσότερα ορυκτά καύσιμα ε, είναι τα πιο καταστροφικά τμήματα, δηλαδή οι δοκότρατες και οι τράτες βυθού. Οπότε η ενίσχυση de minimis έχει δεκαπλασιαστεί ήδη από το 2008. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιχορήγηση προς τον κλάδο αυτό ταυτόχρονα ε, στη διεθνή σκηνή έχουμε ήδη δώσει πολλέ υποσχέσει να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, παραδείγματο χάρη, από 80 έω 95% μέχρι το 2050. Υποσχεθήκαμε επίσης ε, να καταργήσουμε τις ε, ε ουσίες που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον στην Αγκόγη. Αυτό μέχρι το 2020, τα πλαίσια του ΠΟΕ ασχολούμαστε με τον τρόπο μείωση των ενισχύσεων που στρεβλώνουν ε, την ε, αλία. Πιστεύω ότι αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει αυξημένη ενίσχυση minimis τώρα θα υπονομεύσει κατά πάσα πιθανότητα τον ηγετικό ρόλο που έχουμε στις προϊούσες διαπραγματεύσεις ε, περνώντας ένα μήνυμα ανά τον κόσμο ότι και άλλες χώρες ε, μπορούν να αυξήσουν τις επιχορηγήσεις τους για τα καύσιμα στον τομέα της αλίας. Αυτό όμως θα μας οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο και θα αυξηθεί η πίεση που ασκείται στα αλληλευτικά αποθέματα παγκοσμίω και πραγματικά δεν το χρειαζόμαστε αυτό αυτή τη στιγμή, να αναστρέψουμε την τάση. Αυτό χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να περάσουμε πλημελή μηνύματα. Η αγορά πρέπει να απορροφήσει την αύξηση των τιμών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού πρέπει να εστιάσει στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την νέα και πολιτική. Σας ευχαριστούμε κυρία Λεύιν. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, η Κομισιόν γνωρίζει την ε, ισχύουσα κατάσταση στον τομέα τη αλληλείας. Οι τιμέ των καυσίμων είναι το ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το μόνο ο μόνος, το μόνο αίτιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αναφερόμενοι στις τιμές των καυσίμων, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η Κομισιόν ενθαρρύνει τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό Ταμείο. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές μας. Μέχρι στιγμής τα κρατη έχουν χρησιμοποιήσει λιγότερο από το 20% του διαθέσιμου κονδυλίου. Οι υψηλέ τιμέ των καυσίμων θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω τη χρήση των μέσων του Αλληλευτικού Ταμείου που βοηθούν στην αναδιάρθρωση του αλληλευτικού στόλου και προσθέτουν περισσότερη αξία στα αλληλευτικά προϊόντα, βελτιώνοντα έτσι τις τιμές. Είναι πιθανό πως οι τιμέ των καυσίμων θα παραμείνουν ψηλά στα επόμενα χρόνια. Ε, φυσικά την περασμένη εβδομάδα οι τιμές έπεσαν λίγο. Όμως ε, μπορούμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν ε, σκέφτεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινή ελευτικής πολιτικής και του δημοσιονομικού κανονισμού πώς να παροτρύνει για αλληλεία που χρησιμοποιεί λιγότερο τα εντατικά τα καύσιμα. Στόχος θα είναι να ενθαρρυνθεί η προσαρμογή του τομέα και να μπορέσει έτσι να αντιμετωπίσει καλύτερα τις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να σέβεται την αρχή ότι οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια μπορεί δεν μπορεί μάλλον υπό καμία προϋπόθεση να αυξήσει την αλληλευτική προσπάθεια. Στόχος θα είναι επίσης να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα τα λιευτικά θα είναι σύμφωνα με την ε, μάξιμο, με την μέγιστη ε, αλλιευτική δυνατότητα. Περισσότερα ψάρια σημαίνει περισσότερες ελευτικές ε, ε, ε, δυνατότητες και αυτό σημαίνει ψηλότερα εισοδήματα για ολόκληρο τον τομέα. Όσον αφορά την αύξηση του de minimis, της de οροφής, αυτό δεν είναι νέο θέμα. Η Κομισιόν έχει διεξάγει σχετική μελέτη το 2008, αναλύοντας τις επιπτώσεις της μετακίνησης από την οροφή των 3.000 ευρώ στις 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Καταλήγει η μελέτη στο πόρισμα ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την πρόταση για τους εξής λόγους. Καταρχήν μια τέτοια αύξηση θα στρέβλωνε τις αλληλευτικές ε, δραστηριότητες ε, ε, προς περισσότερο εντατικές ε, τεχνολογίες όσον αφορά τα καύσιμα, ε, βλάπτοντας έτσι ακόμη περισσότερο το θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, λιγότερα λευτικά σκάφη, τα ε, μάλλον λιγότερα μεγάλα λευτικά σκάφη θα έπαιρναν μεγαλύτερη επιδότηση και βοήθεια από ό,τι τα μικρότερα. Εμείς δεν θέλουμε να θαρρύνουμε τα μεγάλα σκάφη, ώστε να χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο καύσιμα, αντίθετα. Και τρίτο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Και εδώ το τρίτο θέμα είναι ότι το πολλά κράτη-μέλη ε, είναι αναγκασμένα να επιβάλλουν μέτρα λιτότητες. Και γι' αυτό θα υπήρχαν μόνο θα υπήρχε πολύ περιορισμένη πολιτική στήριξη από τα κράτη-μέλη για μια πρόταση που θα οδηγούσε σε αύξηση των δημοσίων δαπανών. Ακόμα και αν το όριο de minimis αυξανόταν, πολλά κράτη-μέλη δεν θα είχαν τα χρήματα για να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα δυνατότητα για να δαπανίσουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Αν λοιπόν Κάποια κράτη-μέλη μπορούσαν να πληρώσουν ε, μεγαλύτερες ενισχύσεις δεμήνυμης. Αυτό θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό και θα οδηγούσε σε άνισο πεδίο για του αλευτικού στόλου των κρατών μελών. Και αυτό είπαμε είναι πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την εξαίρεση, την φορολογική των καυσίμων για τον αλευτικό τομέα, πράγμα πρότειναν οι πράσινοι, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπιστεί μόνο με νομοθεσία, αλλά πρέπει να συζητηθεί σε σφαιρικό επίπεδο. Η φορολόγηση των καυσίμων που γίνεται μόνο στα ευρωπαϊκά λιμάνια θα οδηγούσε σε μαζικέ ε, ανταγωνιστικές στρεβλώσεις ε, προς ε, ζημία των ευρωπαϊκών στόλων. Επίσης, θα οδηγούνταν πολλά ευρωπαϊκά σκάφη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό και καλούμε τα κρατημένα να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά του λευτικού Ταμείου. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές που έχουν εγγραφεί εξ ονόματος των ομάδων ξεκινώντας από τη συνάδελφο Φράγα Εστέβες. Πρόεδρε, Αναμένοντα τι προτάσει για, για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, το ΕΛΚ θέλει να καταδείξει για άλλη μία φορά την ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση που διανύει ο αλληλευτικό τομέα. Μέχρι ότου υπάρξει μια νέα πρόταση για την κοινή οργάνωση των αγορών σε αυτόν τον τομέα, ο τομέα αυτό ε, έχει μηδενικό περιθώριο όσον αφορά τι τιμέ. Το καθεστώ εισαγωγών πολλές φορές από παράνομη αλληλεία είναι μια στρέβλωση του ανταγωνισμού οι ε, υποχρεώσεις ελέγχου απαιτούν μεγαλύτερη κινητοποίηση των, ε, του δυναμικού από πλευρά ε, των επιχειρήσεων και η μεγαλύτερη κρίση δεν ευνοεί ακριβώς τη μεγαλύτερη κατανάλωση ποιοτικών προϊόντων. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε και μια νέα πτυχή όσον αφορά την αύξηση των καυσίμων που πάλι απειλεί για άλλη μια φορά τις επιχειρήσεις προβλέπονται μεταρρυθμίσεις σε βάθο για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Με αυτό το πανόραμα ω κοινικό, πολλέ επιχειρήσει θα έχουν ανάγκη να έχουν ρευστό στη διάθεσή του για να αντιμετωπίσουν τι προσαρμογέ μέσα σε ένα πλαίσιο υποστήριξη που είναι όλο και πιο μειωμένο. Γι' αυτό ε, αυτή η ε, ερώτηση και αυτή η πρόταση ψηφίσματος ε, σε σχέση με την Ευρωβουλή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι υποστηρίξεις δεν έχουν καμία επιβάνηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και επιπλέον η αύξηση των ενισχύσεων που ζητείτε είναι πολύ πιο κάτω από την βοήθεια de minimis προς αυτό τον τομέα σε σχέση με τον τομέα των μεταφορών ή την γεωργία. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπως το 2008 όπου συζητούσαμε τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε την τελευταία στιγμή να υιοθετηθούν. Θέλω να πω ένα πράγμα προς την κυρία Επίτροπο. Αληθεύει ότι κάποια κράτη-μέλη μπορεί να δίνουν ή να μην δώσουν αυτές τις ε, υποστηρίξεις και θα υπάρξει μια διαφορά όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Όμως μεγαλύτερη στρέβλωση για τον ανταγωνισμό είναι εκείνη η οποία απορρέει από την μη χρηματοδότηση του τομέα της αλίας από κάποια κράτη και γι' αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ κυρία Φράγαστερες. Η κυρία Τροτμάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι αλληλείς μας έχουν ενημερώσει για τις ε, συνεχώς αυξούμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ένα πλαίσιο δύσκολο για αυτούς, εξόδου από τους στόλους, μείωση των ποσοστώσεων και έχουμε και την τρομερή άνοδο, την έκρηξη των ε, τιμών του πετρελαίου. Βέβαια τελευταία έχει λίγο μειωθεί αλλά κυμαίνεται ε, απότομα και αυτό εδώ και δύο χρόνια επιβαρύνει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων αλλιέων ιδιαίτερα την ε, βιοτεχνική και παράκτη αλληλεία. Η κατάσταση είναι ανισχυτική. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, σταθούμε αλληλέγγυοι προς τους αλείς. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να αυξήσει τις βοήθειες de που μπορεί να δοθούν στους αλείς για να αντιμετωπίσουν τα της κρίσεως. Πρόκειται για ένα μεταβατικό μέτρο, αιτιολογημένο από το κοτεπήγον του προβλήματος. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντιδράσει μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο και με μπροστά σε μια τέτοια νέα κορύφωση θα πρέπει να δράσουμε. Να μας πει η Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει. Όπως είπε και η κυρία Φράγκα Εστέβες, είναι σημαντικό να επαληθεύσουμε ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το σύνολο των ποσών που προβλέπονται από τον κανονισμό τα πλαίσια της νέας αλληλευτικής πολιτικής φαίνεται να καθορίζονται πλέον. Διαπιστώνουμε ότι οι αλληλείς δεν είναι πολύ διστακτικοί για τις αλλαγές αυτές. Αντίθετα κάποιοι έχουν ξεκινήσει να κάνουν προσπάθειες για την διατήρηση των αλλιευμάτων είναι μια συλλογική ευθύνη αυτό θα έλεγα. Για να γίνει αυτό δεν θα πρέπει να πέφτουν θύματα εξωτερικών παραγόντων επί των οποίων δεν έχουν καμία δυνατότητα επιρροής. Μια ταχυτάτη απάντηση από πλευρά σας κύριε Επίτροπε θα ήταν ένα μήνυμα το οποίο θα συνεισφέρει τα μάλλα στη σύσφυξη των δεσμών που ιστορικά έχουμε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο συγκεκριμένο, ε, στην συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Ο κύριος Ντέιβις για 1,5 λεπτό. Σήμερα, λόγω της αύξησης των τιμών έχουμε την έκκληση των αλλιέων. Αύριο θα έχουμε τους, γεωργείς, τους γεωργούς, συγγνώμη, μεθαύριο τους ιδιοκτήτες αεροπορικών επιχειρήσεων. Στο τέλος και αυτοί που πολλούν βενζίνη στο δρόμο θα διαμαρτύρονται λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Νομίζω ότι αυτή είναι απαράδεκτη πολιτική στήριξη συγκεκριμένων συμφερόντων αμερικανικού τύπου όπως το κάνουν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Όλοι λένε ότι πρέπει να έχουμε αηφόρες πολιτικές στην αλληλεία. Στην ουσία όταν φτάνουμε στο ψαχνό κανένας δεν καταλαβαίνει τι θα πει αηφορία. Κανένας δεν μπορεί να πει ποιο είναι το νόημα αυτής της λέξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι κατανοεί ότι δεν είναι βιώσιμη η αλλιευτική δραστηριότητα σε ορισμένες τις μορφές, όχι όμως λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, αλλά λόγω ακριβώς κάποιων απαράδεκτων αλλιευτικών πρακτικών επί δεκαετίες. Αν δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μπορέσουν το κόστος το επιπλέον να το περάσουν στους καταναλωτές τους, τότε θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην τιμή των καυσίμων και στο κόστος του προϊόντος. Αλλά το να υποστηρίζουμε μία ή φόρες πρακτικές δεν είναι τρόπος και δεν θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του παρελθόντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε πει στην αρμόδια δική μας Επιτροπή ότι ε, δεν ήταν στόχος της να υπάρξουν επιδοτήσεις για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους των καυσίμων και χαίρομαι ε, που το ξαναείπε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Ντέιβις. Ο κύριος Γκρόμπαρτσικ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η κοινή αντιευτική πολιτική με βάση την αρχή της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να προστατεύει και να διασφαλίζει την διαχείριση των ευρωπαϊκών αλλιευμάτων με ένα ισόρροπο τρόπο. Υπό αυτό το πρίσμα οι αλλιείες και τα, η αλλιεία και τα αλλιεύματα έχουν ζωτικό χαρακτήρα. Όμως η αλλιεία είναι και η μεταφορά διαφανών αξιών από τη μία γενεά στην άλλη, η μεταλαμπάδευση αυτή αυτών των αξιών υπό οικονομικό πρίσμα είναι θεμελιώδους σημασίας να διατηρήσουμε την οικονομική ισορροπία πραγμάτων και δεδομένων των αυξήσεων που είναι δραστικές συστημές των καυσίμων στην Ευρώπη η κοινή αλλιευτική πολιτική θα έπρεπε να εξοπλιστεί με ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει στους αλείς να μπορούν να προστατευθούν από τέτοιου ε, εκρηκτικού τύπου αυξήσει τιμών καυσίμων. Μετά τα προβλήματα των αναπηγείων και των ε, ναυτιλιακών μεταφορών δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει κι άλλον ένα ε, τομέα που αφορά τη θάλασσα και μάλιστα υπέρ της από Ανατολής. Και βλέπουμε, αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο διστάζει η Ισλανδία να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία λοιπόν μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτική πολιτική πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να διασφαλίσουμε ότι το φυσικό περιβάλλον θα προστατεύεται και επίση θα προστατεύονται και οι αλληλεί εξίσου. Για άλλη μία φορά βλέπουμε πάλι το ότι αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της περιφερειοποίησης ε, της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, και δίνεται ιδιαίτερος, ε, μεγαλύτερος ρόλος στις κυβερνήσεις στην αλλιευτική πολιτική και πάλι. Επαναλαμβάνω, δεδομένης της κρίσης ως συγκυρίας και της αστάθειας των πραγμάτων, πάβει ή σταματά να λειτουργεί η κοινή αλληλευτική αλλιευτικη πολιτικη και θα αφήσει τους αλλοί στη μοίρα του. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οφείλω να πω ότι με ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό η απάντηση της Επιτρόπου κυρίας Δαμανάκη για την ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του πετρελαίου για τους αλληλείς. Βρισκόμαστε ενώπιον ε, ενό ζητήματος ε, συνέπειας, αν θέλετε, τη πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωση, Διαρθρωτικός πώς είναι βαριά η τάση, δηλαδή η αύξηση της τιμή ε, του πετρελαίου που ξέρουμε ότι θα διαρκέσει και ότι δεν σχετίζεται μόνο με τα όσα διαμείβονται τώρα στη Βόρεια Αφρική. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μην δώσουμε συγκυριακή απάντηση, δηλαδή αύξηση των επιχορηγήσεων ε, λόγω των διακυμάνσεων που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή ε, στη, στη, στην τιμή του πετρελαίου. Είναι θέμα λογικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δείξει συνέπεια σε σχέση με τους προσδιορισμένους στόχους της, ε, δηλαδή καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών που συνιστά προτεραιότητα, καθώς και μείωση των εκπομπών ε, των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Είναι σημαντικό να μην στείλουμε αντίστροφα διαφορετικά μηνύματα και να μην έχουμε αντιφατική πολιτική. Ε, δεν πρέπει να δράσουμε με τρόπο ώστε να συνεχιστεί ένα ήδη καταδικασμένο ε, ενεργειακό πρόγραμμα για τους αλληλείς. Ε, δηλαδή θα πρέπει να τους αφήσουμε να ανακυκλώσουν ε, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και να διαθέσουμε τα παραγωγικά τους μέσα σε τομείς που μπορεί να είναι βιώσιμοι. Δηλαδή τις επιχορηγήσεις μας θα πρέπει να τις προσανατολίζουμε προς αυτό και όχι να λειτουργούν συγκυριακά για να απαντήσουμε στην τωρινή διακύμαση τιμή του πετρελαίου. Σας ευχαριστώ ευχαριστούμε. Και τώρα θα περάσουμε στους λοιπούς ομιλητές. Ο κύριος Βαλέσα για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε ήδη το 2008 Τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τους ε, προς και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέτρων που θα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαμβληθούν τα πλήγματα για τις περιφέρειες ε, στις περιφέρειες που εμπλέκονται ιδιαίτερα στο έργο της αλίας. Τριπλάσια ήταν η αύξηση του κόστους ε, όσον αφορά την αλία από το 2003 σήμερα τώρα πρέπει 40% να επενδύουν μεγαλύτερα ποσά οι αλληλείς ώστε να μπορούν να καταφέρουν να αλλιεύουν και να διοχετεύουν τα αλλιεύματά τους στους ε, καταναλωτές. Και αυτό σαν αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών καυσίμων. Η οικονομική κρίση είναι κυρίως υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση των πραγμάτων. Και δεδομένου το ότι τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρες ε, diesel, αύξηση των καυσίμων αυτών είναι ιδιαίτερα επώδυνη στους αλείς που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους σκάφη και κινητήρες. Όλο και περισσότερο πρέπει να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις οι αλείς ε, για να αλλιεύουν και αυτό σημαίνει κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας, μεγαλύτερου όγκου καυσίμων. Και η υποστήριξη στο πλαίσιο de minimis θα πρέπει να αυξηθεί από 30.000 σε 60.000 ευρώ και μάλιστα για μια περίοδο τριετή. Αυτό θα βοηθούσε εκείνους ε, που ασχολούνται με την αλία και που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και θα άξανα και την ανάπτυξη την οικονομική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άνδρες Παρέα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το γεγονός ότι σε αυτή την Ολομέλεια που έχει υπερφορτωμένη ημερήσια διάταξη βρήκαμε ένα κενό χρόνου για να συζητήσουμε αυτό το θέμα αποδεικνύει τη σημασία που δίνει σε αυτό το θέμα η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η σημασία, η σπουδαιότητα του τομέα τη Είχαμε μεγάλη αύξηση του βαρελιού πετρελαίου. Αληθεύει ότι σήμερα μειώθηκαν οι τιμέ, όμω παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα αηφορία. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστέ ανησυχούμε για αυτή την κρίση που πλήττει τον τομέα τη αλεία και είμαστε πεισμένοι ότι η λύση βρίσκεται σε μια κοινοτική απάντηση που θα λαμβάνει υπόψη αυτά τα θέματα που πάντα ζητούσαν να ληφθούν υπόψη οι ευρωβουλευτέ ε, και να ληφθούν υπόψη και από τι κυβερνήσει. Ζητούμε να ληφθεί υπόψη η ανάγκη δεδομένη αυτή τη κατάσταση μέσω ενό δίκαιου, σωστού, αποτελεσματικού μηχανισμού να προβλέψουμε κατεπήγοντα μέτρα στο κοινοτικό επίπεδο. Το 2007 εγκρίθηκαν τα μέτρα de minimis. Δεν ζητάμε μόνο τα μέτρα de minimis που θέλουμε να εξεταστούν. Ζητούμε από την Επίτροπο Δαμανά να εξετάσει το άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Αλία που θα δώσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο να δράσουμε γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να δράσουμε χωρίς να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ε, δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει νέους τρόπους προσέγγισης και δράσης ώστε από το Κοινοτικό Ταμείο Αλληλείας να κινητοποιηθούν τα κονδύλια ώστε η, η ε, βιοτεχνική αλληλεία, οι ε, αλληλείς εκείνοι οι οποίοι καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις να μπορέσουν να βοηθηθούν. Να μελετήσετε τη δυνατότητα για την κοινή αλληλευτική πολιτική νέων μέτρων κυρία Επίτροπε, μέτρων που θα ενισχύσουν ε, την ε, δυνατότητα δράσης ε, των αλλιέων σε σχέση με τις τιμές καυσίμων και θα βελτιώσει και την εμπορευματοποίηση των προϊόντων. Όλα αυτά υπό το πρίσμα της αηφορίας που είπατε και της βιωσιμότητας κοινοτική, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής. Αλλά να δούμε και τον ανθρωπιστικό τομέα. Ε, υφίστανται τα πάνδυνα οι αλλιείς. Θεωρούμε ότι είναι ένα κατεπήγον μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ένα μέτρο προσωρινής ελαστικότητας που θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα σε αυτό τον τομέα που πλήττεται τόσο έντονα. Ευχαριστώ. Μπιλμπάο Μπαραντίκα παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αναγκαία μέτρα κατεπήγοντα και συγκεκριμένα για να μειωθεί η επίπτωση που έχει στον αλληλευτικό τομέα η αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ο τομέα εργάζεται με αλλιεύματα που είναι όλο και πιο ε, σπάνια. Έχει όλο και λιγότερε, χαμηλότερες τιμές για αυτά τα προϊόντα και έχουμε και στρέβλωση τη αγορά από τα εισαγόμενα προϊόντα από άλλε χώρε. Ε, υποστηρίζουμε τα αναγκαία αποτελεσματικά μέτρα που δεν θα επιβαρύνουν το κόστος των ευρωπαϊκών προπολογισμών. Όμω, μια και εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα αυτό ο τομέα και δεδομένη τη νέα μεταρρύθμιση κοινή αλλιευτική πολιτική, πέρα από τι προσπάθειε που έγιναν μέχρι τώρα, θα πρέπει να ληφθούν να γίνουν προσπάθειες για μια πολιτική καινοτομία για να βελτιώσουμε με αυτόν τον τρόπο ενεργειακά τον αλλιευτικό στόλο. Διότι το να υποστηρίξουμε αυτή τη δράση είναι και ένα στίχημα υπέρ της αηφορίας. Μια ευκαιρία για την ναυπηγική δραστηριοποίηση και για τον ενεργειακό τομέα για να υπάρξει ένα μέλλον και να μπορέσει να συνεχίσει ο τομέας αυτός τη δράση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Νικουλέσκου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, είναι λοιπόν πραγματικά πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε το ότι δεν θα έχουμε ποτέ ξανά επίπεδα 30-40 δολαρίων για το ε, αναβαρελί. Δεν θα υπάρξουν πια τέτοιε τιμέ ε, πετρελαίου. Θα πρέπει να υπολογίζουμε με τουλάχιστον 80 δολάρια το βαρέλι. Και θα έχουμε τι αρνητικέ επιπτώσει που θα συνεχίζονται λόγω τη αύξηση των καυσίμων. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα σε ευρωπαϊκό τομέα. Οι Ευρωπαίοι αλληλεί αντιμετωπίζουν μια πολύ ένα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό παγκόσμια. Και σε πολλέ περιφέρειε είναι η μόνη η δυνατότητα οικονομική εκεί να επιβιώσουν και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένων των υψηλών τιμών καυσίμων δεδομένων των υψηλών τιμών του πετρελαίου να μην πλήττονται ιδιαίτερα ε, πάντα οι ε, βιοτεχνικοί αλληλείς. Εξαρτάται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αλληλείας ε, από την υποστήριξή τους. Το Ταμείο Αλληλείας θα πρέπει να προσαρμοστεί και να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Κύριος Κρήτον Αρσένης, παρακαλώ, δύο λεπτά. Αγαπητοί Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά δεν θα έχουμε αλία αν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε την ε, κατάρρευση των, των αλλιευμάτων μας, των αποθεμάτων αλίας. Όμως είναι σημαντικό να δούμε και το τι γίνεται στους ε, αλίες μας σήμερα. Και είναι αλήθεια ότι οι μικροί αλίες, οι παράκτη αλίες, είναι αυτοί που υποφέρουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Συντάμε για την διεύρυνση ενός μέτρου στο οποίο είναι αλήθεια ότι στην πράξη λίγες χώρες έχουν πρόσβαση. η οικονομική κρίση θα οδηγήσει τις περισσότερες μεσογειακές χώρες να μην μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το de minimis. αυτό είναι μια πραγματικότητα. από την άλλη θα πρέπει να δούμε πώς μέσα από το κοινό αλληλευτικό μας ταμείο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες που έχουν μια σοβαρή οικονομική κρίση να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα να μπορέσουν να βοηθήσουν τους αλληλείς τους. προσωπικά στηρίζω την ε, διεύρυνση του de με κάποιες προϋποθέσεις. οι προϋποθέσεις είναι να δοθεί έμφαση στους μικρούς αλείς στη μικρή και παράκτια αλεία να δοθεί έμφαση στους αλείς που εφαρμόζουν ορθές βιώσιμες αλληλευτικές πρακτικές να δοθεί έμφαση έτσι ώστε η χρηματοδότηση να μην οδηγεί στην αύξηση της αλληλευτικής προσπάθειας και τα μέτρα αυτά να μην απειλήσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλίας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε να μην αποθαρρυνθεί η ευρωπαϊκή αλία από το να γίνει ενεργειακά πιο αποδοτική. Και Επίτροπε, συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε περισσότερο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, ιδιαίτερα πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν έχουν πλέον τους πόρους να συμμετέχουν με την ίδια συμμετοχή στο να συμμετέχουν πιο ενεργά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αρσένη. Η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε, επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε επιβάλει διάφορους όρους και απαιτήσεις για να είναι βιώσιμη η αλληλευτική μας πολιτική. Ταυτόχρονα όμως οι αλληλείς χρειάστηκε να προσαρμοστούν διότι η αυξημένη τιμή του πετρελαίου είναι αδυσβάσταχτο άχθος για αυτούς. Έχει σχεδόν γονατίσει ο κλάδος. Η αρχή de minimis ε, θα υπάρχει μέχρι το 2013 ως έχει. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την αρχή αυτή de minimis, αν είμαστε ε, σοβαροί σε σχέση με το προσανατολισμό που θέλουμε να δώσουμε στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Οφείλουμε να αναρωτηθούμε το εξή. Επαρκεί η νομοθεσία της Ένωσης για να ε, θωρακίσουμε τα συμφέροντα των ε, στον τομέα της μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο διπλασιασμού του ορίου de minimis από 30.000 σε 60.000. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη ώστε να χρησιμοποιήσουν τους ε, υφιστάμενους πόρους ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας ε, τηρούν σιγή ηχθείως κάποια κράτη-μέλη διότι θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να υπομιστούν άλλο άχθος ε, και παραπέμπουν το θέμα στις Βρυξέλλες. Ε, βέβαια, οι αλληλείς μας, ας πούμε, δεν γνωρίζουν καν ε, τις ε, δυνατότητες που είναι στη διάθεσή τους. Έχουν υποβάλει σχετική ερώτηση στην κυβέρνηση επανειλημμένη, αλλά δεν γνωρίζουν όμως τον κανόνα περί ενισχύσεων de minimis. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβαλούν κάθε δυνατή προσπάθεια τους ώστε να απορροφηθεί από τον κλάδο το χτύπημα της αύξησης τιμής ε, του πετρέλαιου. Είναι θέμα επιβίωσης. Αφήστε που είναι και επαχθέστατη η διαδικασία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και δεν ξέρω από αυτό τον κανόνα για τις ενισχύσεις de Ευχαριστούμε τον κύριο Καντέκ που γύρε το ζήτημα. Και προσθέτω μία επερώτηση. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν ορθότερα τον κανονισμό de και τι θα κάνει η Επιτροπή ούτως ώστε να επιτύχουμε ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο της απορρόφησης των κονδυλίων και τη δυνατότητα απορρόφησης από πλευρά των αλλιών. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η αύξηση των τιμών ε, πετρελαίου είναι μια διαθροτική τάση σε σχέση με την αύξηση της γενικής ζήτησης. Ε, έχουμε την το ευμετάβλητο χαρακτήρα που τα τελευταία ε, χρόνια ε, απέτησε μια προσαρμογή. Πρέπει να περιοριστεί η αύξηση του κόστους όσον αφορά την ε, αλληλεία που πολλές φορές περιπλέκει ιδιαίτερα το μέλλον του, του τομέα της αλληλείας. Όταν γίνεται λόγος για τον τομέα de minimis, εδώ δεν θα πρέπει να ε, χαρκεύεται ο ανταγωνισμός. Πρέπει να αξιολογηθούν αυτές οι πτυχές, αλλά να πάμε σε μια πιο φιλόδοξη λύση που θα λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική για την θάλασσα, τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θεωρώ ότι μια απάντηση συνεκτική και με συνάφεια πρέπει να αυξήσει τη δυνατότητα προσαρμογών, διαθετικών προσαρμογών στην Αλία και να βοηθηθούν οι πιο ευάλωτοι του τομέα. Ιδιαίτερα η μικρομεσαίη παραγωγή και η βιοτεχνική αλληλεία. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, προσέγγιση της Επιτρόπου και την ε, ε, χρήση των κονδυλίων της αλληλείας πρέπει να συνδυαστούν και με μακροπρόθεσμη προσέγγιση για μια μεγαλύτερη αηφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάντζες Πρεσέντο. Στα ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι αλληλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τρει βασικές δυσκολίε. Πρώτον, το θέμα των ποσοστώσεων, περίπλοκο θέμα, τους οδηγεί να υιοθετούν πρακτικές καταναγκαστικέ. θα έλεγα. Δεύτερον, η έλλειψη κατάρτιση, η υποβάθμιση τη δραστηριότητά του. Και τέλος, και αυτό συζητάμε σήμερα, αύξηση των τιμών του πετρελαίου που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την δραστηριότητα αυτή που βρίσκεται πλέον σε βαθιά κρίση. Από το 2008 στο 2010 οι διακυμάνσεις του πετρελαίου οδήγησαν στην απώλεια κάνα εβδομάδα 100 με 200 ευρώ. Αυτά στους Γάλλους και εγώ προέρχομαι από μια αλλιευτική πόλη και γι' αυτό απαιτώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις βοήθειες ντεμίνιμης. Το μέτρο αυτό θα μειώσει τις ποιώσεις που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι αλληλείς για να ζήσουν ε, από την δραστηριότητά τους χωρίς αυτό να επηρεάσει αρνητικά την ανανεώση των αλλιευμάτων. Η μελλοντική αλλιευτική πολιτική πρέπει να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σήμερα την ημέρα της Ευρώπης ακούει τους αλληλείς. Αυτό θα είναι μια καλή αρχή επίτροπε από σας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Κύριος Φερέιρα τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Η σημαντικότατη αύξηση των τιμών των καυσίμων έπληξαν σε σημαντικότατο βαθμό τομεί όπως η αλληλεγγύη. η, η οικονομική βιωσιμότητα έχει πληγεί ε, και λαμβάνουμε υπόψη φυσικά και τα ήδη χαμηλά εισοδήματα των αλίων. Η διακύμανση των τιμών για, όλους τους, ε, για όλα τα παραγωγικά μέσα δεν μπορούν να αντισταθμιστούν πλέον από τον κλάδο και σε αυτό προσθέτουν και άλλο προβλήμα προβλήματα ε, όπως αυτό των εισαγωγών. Ε, εδώ και χρόνια έχω έχει επέλθει σε τέλμα ο κλάδο ε, ή έχουν μειωθεί οι αποδόσει και αυτό μετακυλείται φυσικά και στι τελικέ τιμέ του ε, για τον καταναλωτή. Με τη νέα κοινή ελευτική πολιτική δεν λειτουργήσαμε επαρκώ ικανοποιητικά και δεν κατανείμεται επαρκώ η προστιθέμενη αξία σε όλη την αλυσίδα του κλάδου. Ε, τα τελευταία χρόνια επίσης είδαμε ότι έχουν εκλείψει διάφορες δραστηριότητες και κινδυνεύουν να εκλείψουν εκατοντάδε χιλιάδε εκμεταλλεύσεις ε, και όχι μόνο και παρακτήων πολλών που εξαρτώνται από την αλληλεία και άρα από τι σημαντικέ ε, τιμέ ε, του πετρέλαιου. Σε σημαντικό βαθμό πλήττεται η ρεσταχνική αλληλεία και μην ξεχνάτε ότι σε χώρε όπω η Πορτογαλία το 90% του αλευτικού μα στόλου είναι μικρά σκάφη. Η αδράνεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η άρνησή τη να δεσπίσει τα απαιτούμενα μέτρα θα μα οδηγήσουν στην καταστροφή και σήμερα η Επίτροπο επιβεβαίωσε αυτή τη θέση. Μία λύση μα προτείνεται, Επίτροπε, μόνο για τον στον κλάδο ε, χωρίς καμία διαφεροποίηση να παραπληστούν ουσιαστικά ε, κάποιες, ε, κάποια αλλιευτικά σκάφη. Δηλαδή τι τα βάζουμε με την αρρώστια, την να ασχολούμαστε με τον ίδιο τον άρρωστο και μην ξεχνάτε ότι κάθε χώρα έχει ιδιαιτερότητες, έχει διαφορετικές ανάγκες και τίποτα δεν έχει λυθεί σε ορισμένες χώρες με τα νέα μέτρα της αλλιευτικής πολιτικής. Γιατί όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ευθύ αμέσω να δώσουμε μία ε, ικανοποιητική απάντηση, όπως παραδείγματο χάρη να θεσπίσουμε ένα ταμείο εγγυήσεων όπου όλοι θα συμμετέχουν σε επίπεδο Ένωσης ε, για να εγγυηθούμε τη σταθερότητα των τιμών ε, των καυσίμων. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της Ένωσης για χρηματοδότηση εκτάκτων μέτρων στήριξης του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη όμως της διαρθρωτικής τάσης και της διαρκούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου, οφείλουμε να εξετάσουμε το θέμα Τη βιωσιμότητας της αλίας, ε, την μέσο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου ε, σε διάφορες χώρες. Ε, χρειαζόμαστε μια χαμηλότερη τιμή της πρώτης πώληση και καλύτερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε ολόκληρη την αλυσίδα. Το Ταμείο Αλίας πρέπει να στηρίξει τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών στόλων, να επιλέγονται καλύτερα τα αλλιευτικά μέσα, να θεσπίσουμε τα απαιτούμενα μέτρα για τους κινητήρες των σκαφών για να είμαστε και φιλικοί προ το περιβάλλον και να υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων. Οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκέ απαντήσει, αλλά όχι να διωγγώσουμε τι ανισότητε που ήδη παρατηρούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και που διωγγώνονται λόγω τη βαρύτητα τη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση που ε, πλήττει τι ε, πλέον ευπαθεί οικονομίε. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Αντροβέρ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Η διατύπωση ερώτηση είναι. Σε σχέση με την απάντηση σε αυτή την περίπτωση που μπορεί να θεωρηθεί απογοητευτική απάντηση. Ο τομέα αλληλείας προφανώς βρίσκεται σε κρίση. Το εισόδημα των αλληλείων είναι κάθε φορά μικρότερο και περιπλέκεται η ε, συνέχιση των δραστηριοτήτων. Και δεν κάνουμε λόγο εδώ για συγκαλυμμένες ε, ε, επιχορηγήσεις. Κάνουμε λόγο για πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν και πρέπει να υποστηριχθούν από εμά για μια δίκαια, ε, δίκαια διεκδίκηση αυτού του τομέα. Δεν είναι κάτι το μεμπτό αυτό. Αν το αντίθετο, πρέπει να είμαστε συνεκτικοί. Και εδώ δεν αμφισβητείται ο τομέας αλίας. Γιατί πρέπει να απορριφθούν μέτρα συγκυριακά περιορισμένου έκτακτου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση έκτακτων τέτοιων χαρακτηριστικών θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τομέα που χρειάζεται άμεση βοήθεια και θα μπορούσε να εξεταστεί και η βοήθεια τεμήνυμης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άλμπες. Και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου, Πρόεδρε, σε όλου εκείνου που εδώ εξέφρασαν ανησυχίε σε σχέση με την δραστηριότητα των αλλιέων. Με χαμηλέ τιμέ αλλιευμάτων και υψηλότατε τιμέ καυσίμων, ιδιαίτερα του τελευταίου μήνε. Όπω πολύ καλά αναφέρθηκε, το κόστο των καυσίμων έχει ιδιαίτερε επιπτώσει για την επιβίωση των μικρών αλλιέων και ιδιαίτερα επιδεινώνει την επιβίωσή του με ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτή η αύξηση των ε, καυσίμων έχει ε, βαθύτατε αρνητικέ επιπτώσει. Ε, δημιουργεί μια στενοπόγια του αλληλεί όσον αφορά το εισόδημά του, Με αύξηση των εισαγωγών από τρίτε χώρε και γεωργικών και αλλιευμάτων, γεωργικών προϊόντων και αλλιευμάτων και υπάρχει και εγκατάλειψη του τομέα λόγω δυσκολία και απώλεια θέσεων απασχόληση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κρίση πρέπει να δράσουμε. Να δράσουμε ταχύτερα σε βάθος, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της αλληλεία στη ρίζα τους. Γι' αυτό αναμένουμε θετικές ε, ε, απαντήσεις και ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα με άμεσες ε, δράσεις που θα υιοθετηθούν, ώστε να βοηθηθούν οι αλληλεί μας. Ευχαριστώ. Grazie, collega, la parola. Ευχαριστούμε. Ρωμέβα Ιρουέδα παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να είμαστε σαφείς. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη να υπάρξει αναδιάθρωση στην Αλία, ώστε να μην είναι ε, ενεργοβόρα τα σκάφη και κινητήρες και να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη αηφορία μακροπρόθεσμα και να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα κοινωνικά και οικονομικά. Γι' αυτό το να, δοθεί, να δοθούν μεγαλύτερα κονδύλια στον τομέα της αλληλείας λόγω της αύξησης των καυσίμων θα έστελνε ένα εσφαλμένο μήνυμα κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής και θα έδινε ένα κίνητρο στους ε, ε, πλειοκτήτες να χρησιμοποιούν περισσότερο ενεργοβόρους κινητήρες. Αυτό θα ήταν εσφάλμα και εδώ θα πρέπει να δούμε σε σχέση με το διαθετικό χαρακτήρα τα προβλήματα. Μας δείχνει η συγκυρία ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αλλιευμάτων που δεν αλλιεύεται. Οποιοδήποτε μέτρο λοιπόν θα μπορούσε να υιοθετηθεί σχετικά θα ήταν ένα θετικό μέτρο. Κάνοντας το αντίθετο θα ήταν ένα πολύ αρνητικό μέτρο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Άκουσα δύο συναδέλφους να θέτουν ορισμένα θέματα για το θέμα της αηφορίας και για το ότι θα πρέπει να επιδοτηθεί υποτίθεται ε, η συγκεκριμένη δραστηριότητα γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι αλληλείς αυτό που ζητούν είναι να ζήσουν από τη δουλειά τους, από τον υδρότα τους. Αν το πετρέλαιο είναι ένα συγκυριακό πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει αντίστοιχο πρόβλημα και στο μέλλον και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε την έρευνα να βρει μηχανές εσωτερικής καύσης λιγότερο ενεργοβόρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να μην αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας. Βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση της τιμής του αλλιεύματος για τους αλείς ενώ το σημείο πώληση στη Λιανική η τιμή έχει φτάσει στα ύψη και μόνο οι πλούσιοι αγοράζουν. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μεταρρυθμίσουμε τις ποσοστώσεις αλλά και τις πρακτικές του επαγγέλματος που βοηθάει τους μεγάλους και δεν βοηθάει καθόλου αλλά καταστρέφει τους μικρούς Bones. Bonds. Ευχαριστώ. Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου προσθέτουν προβλήματα στους αλλιείς, αλλά δεν είναι το πρώτο, είναι το τελευταίο πρόβλημα. Για τον Βρετανικό αλλιευτικό στόλο, που είναι ο μεγαλύτερος ίσως, ξέρετε ότι παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 70% των αλλιευμάτων που καταναλώνονται, αλλά δεν έχει δικαιώμα παρά μόνο στο 30% των ποσοστώσεων tonnes before joining what was then the EEC έχουν τα αλλιεύματα τα οποία εκμεταλλεύονται οι Βρετανοί αλληλείς έχουν μειωθεί κατά 30% τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλοί αλληλείς διώκονται από το επάγγελμα. Στο τέλος οι αλληλείς θα θέλαν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά όμως ζητούν καλύτερη και πιο δίκαιη αντιμετώπιση. αυξάνουν τις, ε, τα ωράρια ε, αλληλείας χωρίς αυτό να οδηγεί από τον Βρετανικό στόλο στην υπεραλίευση. Ενώ η υπεραλίευση ασκείται από όλους τους άλλους. Ευχαριστώ συνάδελφε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη. Έχετε το λόγο κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να κατανοήσω όλες τις ανησυχίες σας βέβαια και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας πρέπει να πω για τα χαμηλά εισοδήματα των αλλιών μας, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών μικρών σκαφών και ιδιαίτερα παράκτιων περιοχών. Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέρχεται από την αύξηση των καυσίμων. Είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Συζητήσαμε αυτό το πρόβλημα επανειλημμένα και αναγνωρίσαμε ότι υφίσταται αυτό το πρόβλημα και ότι το είχαμε ακόμα και πριν από την αύξηση καυσίμων. Ακόμα και πριν από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Φυσικά μπορώ να κατανοήσω ότι η αύξηση των τιμών καυσίμων μπορεί να επιδεινώσει, να εντείνει το πρόβλημα. Όμω ο κύριο λόγο, ο κύριο λόγο του προβλήματο είναι όπω πάντα η υπεραλίευση. Η υπεραλίευση η αλίευση πέρα και πάνω από τα όρια <clears throat> που δεν μπορεί και δεν αφήνει τα αλλιεύματα σε υγιή κατάσταση. Αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε με τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλιευτή πολιτική. Τώρα φυσικά συζητάμε για την αύξηση των τιμών καυσίμων. Μάλιστα, αυτό είναι ένα πρόβλημα πράγματι. Και α προσπαθήσουμε να συζητήσουμε το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και μάλιστα μόνιμα και διαρκέστερα είναι να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα του τομέα της αλίας όσον αφορά αυξήσει καυσίμων, αυξήσεις τιμών καυσίμων. Είναι ο μόνος τρόπος αυτός, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη των τιμών καυσίμων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στο Βέλγιο μετά την τελευταία κρίση, μείωσαν και βελτίωσαν σε σχέση με την επίδοση του στόλου τους και τώρα έχουν μία μείωση κατά 20%. 20% μείωση της ε, κατανάλωσης ε, καυσίμων στον αλλιευτικό του στόλο. Αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά όμως, αναφερόμενοι στις προτάσεις σας, πρέπει να πω, υπάρχει μια πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξηθεί το ανώφλι de minimis Ας αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Τι είναι αυτό το ανόφλη. Το ανόφλι τη υποστήριξη που μπορούν να δίνουν τα κράτη-μέλη στον αλληλευτικό τομέα. Τώρα, αν έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυξήσει αυτό το ανόφλη, το, τι θα σημαίνει αυτό. Αυτό θα σημαίνει ότι μόνο εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν υγιεί προπολογισμού μπορούν να παράσχουν τέτοια βοήθεια. Αυτό θα είναι η δημιουργία ενός άνισου πεδίου δράσης και δραστηριοποίησης για τους αλείς. Μόνο για τις πιο πλούσιες χώρες θα μπορεί να λειτουργήσει. Ας το πω αυτό ξεκάθαρα και σταράτα για να γίνει κατανοητό. Ακόμα και να αυξήσουμε το ανόφλι, μόνο τα μεγαλύτερα σκάφη θα μπορούν να υποφεληθούν. Και έτσι πρέπει να πω ότι υπάρχει κάποια έκπληξη να ακούω από μέλη ευρωβουλευτές να κάνουν προτάσεις και να λένε να υπάρξει αύξηση του ανοφλίου. Τα κράτη-μέλη μπορούν τα ίδια να δίνουν τις κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις τους. Και τα πλουσιότερα κράτη-μέλη το κάνουν ήδη τώρα αυτό. Και για τα γεγονότα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Τώρα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μόνο 20% από αυτή τη χρηματοδότηση. Κάποιοι ευρωβουλευτές μου είπαν ότι είναι πρόβλημα αυτή η χρηματοδότηση, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Υπάρχει όμως η ελαστικότητα. Υπάρχει ελαστικότητα και τα κράτη-μέλη μπορούν να αναμεταθέσουν, να αναδιαρθρώσουν τη χρηματοδότηση αυτή. Όλα τα κράτη-μέλη, κάθε κράτος-μέλος μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο η Ιταλία, μόνο η Ιταλία προσέτρεξε σε εμάς και ζήτησε για μια τέτοια μετάθεση και εμείς το εγκρίναμε. Γιατί δεν προσπαθούμε λοιπόν να πείσουμε τα κράτη-μέλη, να πείσετε εσείς τις κυβερνήσεις των χωρών σας να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά με το σωστό τρόπο αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Και αν υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την απορρόφηση των κονδυλίων, να προσέλθετε εδώ, να το αναφέρετε για να, να βοηθηθούν όλοι. Λοιπόν, για να απαντήσω τις παρεμβάσεις και τα ερωτήματα άμεσα. Μάλιστα, η χρηματοδότηση υφίσταται και υπάρχει. Μάλιστα, τα κράτη-μέλη μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα, τα κράτη-μέλη μπορούν και από τις δικέ τους ε, πηγές μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το ανώφλι de minimis. Λοιπόν, το μόνο αποτέλεσμα που θα είχε αν πορευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μόνο τα πλουσιότερα και μεγαλύτερα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να επωφεληθούν και χρησιμοποιώντας και μεγαλύτερα σκάφη. Φυσικά υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά και μπορούμε να το συζητήσουμε σε σχέση με τη μεταρρύθμιση για την αλληλεία. Να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη μικρή κλίμακα αλληλεία, την βιοτεχνική αλληλεία ιδιαίτερα και να συζητήσουμε και όλες τις άλλες προτάσεις, κάθε μια ξεχωριστά αλλά αυτή η πρόταση να αυξηθεί το ανώφλιντε μήνυμης είναι μια πρόταση που δεν θα βοηθήσει και είναι λανθασμένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Τέλος της συζήτησης. Η ψηφοφορία θα γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι. Διακόπτουμε για τρία λεπτά.